θα γίνει αύριο. Προχωρούμε τώρα στις ε, παρεμβάσεις ε, του ενός λεπτού βάσει του 163 του κανονισμού. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ρόλα. Ευχαριστώ πρόεδρε αποφασίζοντας να κλείσει το εργοστάσιο του στον Κόσλι στο Βελγίο, η κατεπηρέ δημιούργησε ένα κοινωνικό σεισμό. Πάνω από 2.000 άμεσε θέσει εργασία άνω των 6 έμεσε. Η απόφαση αυτή είναι απαράδεκτη, πόσο μάλλον που γίνεται παραγνωρίζοντα πλήρω τα δικαιώματα των ε, μισθωτών αλλά και τις θέσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Το 2013 η αλλά δηλαδή, είχε ε, καταργήσει 1.200 θέσεις εργασίας. Ε, οι μισθωτοί και τα συνδικάτα ωστόσο έδειξαν μεγάλη ευθύνη τότε για να διασωθεί η δραστηριότητα της βιομηχανία εκεί με πολλέ παραχωρήσει. Αντί για ευχαριστίε, ε, διώχονται με μια διοίκηση από τις ΗΠΑ που δεν έχει καν το θάρρος να εξηγήσει γιατί το έκανε και που αγνοεί τους βασικού κανόνε του κοινωνικού διαλόγου. Τούτο απαιτεί ταχεία αντίδραση που θα υποστηρίξει και τους εργαζόμενους, αλλά και όχι μόνο, εφαρμόζοντας μια ουσιαστική ε, φιλόδοξη βιομηχανική πολιτική προς όφελος των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Κύριε Νταντσίλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι γυναίκες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον χώρο της υπαίθρου, αντιμετωπίζουν πάμπολες δυσκολίες όταν προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας και απασχόλησης και να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο σταθερότητας για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε τις συνθήκες αυτές ε, που ισχύουν για αυτές τις γυναίκες έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ευημερία, στην, ε, ε, στις οικογένειες, τέτοιες καταστάσεις. Στη Ρουμανία υπήρξε και μια πρόταση λήψης δημόσιων μέτρων, πολιτικών μέτρων που θα έπρεπε να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Διευκολύνσεις για τις γυναίκες στην Ήπεθρο ώστε να μπορέσουν να βρουν μια σταθερή απασχόληση. Υποστήριξη για τις γυναίκες που εργάζονται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και με δωρεάν ε, ελέγχους ε, για το αν είναι έγκαιες ή όχι αυτές οι γυναίκες ε, όταν χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών για τις οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι ηθικά παράδεκτη και πολιτικά εντελώς προκατηλημένη αποτελεί όνειδος για την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση που νύπτει τα σχήρα τη σαν νέος πόντιος πιλάτος στο ζήτημα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων. αποτελεί ταμή ιστορική πρόκληση προς τους έλληνες αγωνιστές της εθνικής αντίστασης αλλά και στους λαούς της ευρώπης που δεν έσκυψαν το κεφάλι στο ναζιστικό θηρίο. αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η ευρωπαϊκή ένωση έχει πλέον μετατραπεί σε γερμανική ευρώπη ακόμη και την ίδια την ιστορία αποτελεί απόφαση που αποθρασύνει ακόμη περισσότερο το βερολίνο όπως φάνηκε από τις σημερινές προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου της γερμανικής καγκελαρίας στέφεν Ζάιμπερτ που δηλώνει ότι το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων έχει δήθεν ρυθμιστεί. Βέβαια η Κομισιόν και οι διάφορες μνημονιακές δυνάμεις στην Ευρωβουλή ενθαρρύνθηκαν από την προκλητική αδιαφορία που έδειξε η κυβέρνηση Τσίπρα που δεν υποστήριξε την αναφορά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ΠΕΑΔΕΣ ΔΟΣΟΕ όμως δεν πρόκειται να το βάλουμε κάτω. ο αγώνας για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων συνεχίζεται. ευχαριστώ. Σελίμοβιτς, ένα λεπτό. Με μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Οι επερχόμενες εκλογές στη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα οδήγησε την, ε, στην, ε, στο σταγματικό των ψήφισμα παρότι το ανώτατο δικαστήριο της Βοσνίας ε, τόνισε ότι αυτό παραβιάζει το κοσμικό σύνταγμα της χώρας ε, το να παίζουμε με τέτοιες προεκλογικές μεθόδους στην Βοσνία είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το δημοψήφισμα δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο την ε, κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας, αλλά μπορεί να γεννήσει νέες συγκρούσεις. Δεν θα πρέπει να ανάψει η αποθήκη της Βοσνίας εκ νέου. Δεν αξίζει η... μια εκλογή την ε, ειρήνη. Γι' αυτό πρέπει να αναλάβει δράση η Ένωση. Αλλιώς η αστάθεια μπορεί να εξελιχθεί και δεν μπορούμε να ζητήσουμε από κανένα να κάνει μια προσπάθεια ειρήνευση. Η Ένωση πρέπει να ζητήσει αμέσως να διακοπεί αυτό το παράνομο δημοψήφισμα. Κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στην Πορτογαλία η οδός της επιστροφής ε, δικαιωμάτων προς τους ε, εργαζόμενους και συνταξιούχους ε, αφορά μία από τις πτυχές τις πιο αρνητικές της προηγούμενης κυβέρνησης και παρότι είναι η ανεπαρκής αυτή η οδός συγκρούεται με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι θέλουν να υπονομεύσουν οποιαδήποτε πολιτική που αμφισβητεί τις, τις τις πριτανεύουσες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι, αυτό είναι το νόημα της αφόρητης κατάστασης επιβολής κυρώσεων εις βάρος της Πορτογαλίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα κονδύλια και την διάθεσή τους με την διαμόρφωση του προϋπολογισμού, κρατικού προϋπολογισμού. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Καθιστά ακόμα πιο καθαρή και ε, φανερή την ανάγκη ρήξης με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το Ευρωπαϊκό Νόμισμα, την, κρατική, την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Πρέπει οι ανάγκες των χωρών να λαμβάνονται υπόψη ε, πέρα από τις ε, διαπραγματεύσεις ε, για το χρέος. Ευχαριστώ. Κύριο Σεμπαστιά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντο τη Ισπανία ε, διαβεβαιώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ούτω ώστε περιοχέ εξαιρέσει προστασία στη Μεσόγειο να, προχω... να ξεκινήσουν εργασίε για την ε, έρευνα, υποθαλάσσια έρευνα για Και Ωστόσο, η κυβέρνηση δίνει άδειε, συνεχίζει παρότι η Επιτροπή διαμαρτύρεται γι' αυτό η κυβέρνηση λέει ότι προστατεύει το περιβάλλον αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει δράσεις που επιβαρύνουν το περιβάλλον και τον τουρισμό που είναι η βάση της οικονομίας της περιοχής. Η Επιτροπή έχει την καταγγελία στα χέρια της της πλατφόρμας των πολιτών που καταγγέλει την κυβέρνηση της Ισπανίας ε, ότι οι άδειε που έδωσε δεν τηρούν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ωστόσο η Κομισιόν σιωπή. Ας ακούσει η Κομισιόν την άποψη των πολιτών και των επιστημόνων που και ας ε, απαιτήσει να, διακοπούν η, να διακοπεί η χορήγηση των αδειών. Ο κύριος Κοράου. <clears throat> Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στη δική μου περιφέρεια, στη Σικηλία, λείπουν περίπου 50.000 εκτάρια φυτών που είχαν την δυνατότητα παραγωγής θέσεων εργασίας, υπεραξίας, οξυγόνου και κυρίως αυτά εδώ που βλέπετε τα λεμόνια. Εμείς έχουμε υπεψηφίσει βέβαια την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με το Μαρόκο που χωρίς να αναγνωρίζει την ανάγκη ε, ελεγχόμενης ετικετοθεσίας και ε, ηχνηλασιμότητας του προϊόντος ε, εισάγουμε πραγματικά προϊόντα που δεν έχουν σχέση με το πραγματικό άρωμα ενός λεμονιού από τη Σικελία. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν λύσεις εδώ και μία δεκαετία. Έχουμε μιλήσει για τις τροποποιήσεις της οδηγίας για την ιχνηλασιμότητα υπάρχουν ρήτρε προστασίας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει, αλλά δυστυχώς τώρα είναι αργά. Ο κύριος Μποργέζιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποιες εβδομάδες πριν ξέρετε ότι ένας τρομερός σεισμός χτύπησε τρεις μεγάλες περιοχές της χώρας μου. Τρεις περιοχές της χώρας μου. Πριν λίγο άκουγα έναν μαχητικό δήμαρχο ε, από ένα από τα κατεστραμμένα χωριά, το Αματρίτσε, και με ρώτησε θα μπορούσε να πάρει το λόγο εδώ, στην Ολομέλεια. Μιας και θα πάει στις ζώνες αυτές μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να μιλήσει η αντιπροσωπεία απευθείας με τους δημάρχους, γιατί εμείς εκπροσωπούμε τον πληθυσμό. Οι πληθυσμοί αυτοί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την περιοχή που ζουν, σίγουρα έχουν ένα πολύ άσχημο χειμώνα μπροστά τους, θέλουν βοήθεια για να συνεχίσουν να εργάζονται, να συνεχίσουν να παράγουν, είναι πληθυσμοί δεμένοι με την περιφέρειά τους και θέλουν να προσπαθήσουν να σώσουν τις περιοχές τους, να σώσουν την ταυτότητά τους. Πρέπει να κάνει η Ευρώπη ό,τι μπορεί το ταχύτερο δυνατόν πρόσφατα η επιτροπή αναφορών του ευρωκοινοβουλίου προσβάλλοντας τα χιλιάδες θύματα της ναζιστικής στηριοδία στην ελλάδα απέρριψε αναφορά της πανελλήνιας ένωσης αγωνιστών εθνικής αντίστασης δημοκρατικού στρατού ελλάδας εκπρόσωποι των οποίων βρίσκονται εδώ στο στρασβούργο για να δώσουν αύριο συνέντευξη τύπου για τη συνεχιζόμενη για δεκαετίες προκλητική άρνηση των γερμανικών κυβερνήσεων για καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τα ναζιστικά εγκλήματα παραβιάζοντας τη διεθνή συμφωνία των παρισίων περί πολεμικών επανορθώσεων που μόνο η ελλάδα δεν έλαβε παρά το ότι αναλογικά είχε τα περισσότερα θύματα. 71 χρόνια μετά την αντιφασιστική νίκη των λαών αντικειμενικά καταδικάζονται πάλι τα θύματα αθωώνονται οι σφαγείς. Μόνο η ευτυχείς η χρυσή αυγή και η άλλη νοσταλγή του χίτλερ. παρά τις μεγαλοστομίες η απαράδεκτη προκλητική άρνηση των ελληνικών κυβερνήσεων και τη σημερινή σύριζα ανέλ να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις υπηρετώντας τις διεθνείς συμμαχίες της ελληνικής αγκιστικής τάξης ενισχύει τη γερμανική αδιαλαξία. το κκε θα κλιμακώσει τον αγώνα του για αυτή τη δίκαιη λαϊκή απέτηση σαν αιμοδότης και πρωτομάχος της εθνικής αντίστασης. Πρόεδρε, Πρόεδρε, η Επιτροπή το Δεκέμβριο πέρυσι υιοθέτησε το πρόγραμμα απελευθέρωσης των θεωρήσεων με την Ουκρανία, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους ε, στην Ευρώπη. Παρότι εκατοντάδες ε, χιλιάδες ε, παράτυπων μεταναστών συνεχίζουν να φτάνουν στην Ευρώπη χωρίς ελέγχους, οι Ουκρανοί μεταξύ των οποίων και οι Ούγγροι της υποκαθπαθικής Ρουθινίας συνεχίζουν να, να, να, ε, χρειάζεται να υποβάλουν θεωρήσεις. Οι Ουκρανοί έκαναν πολλές θυσίε ε, για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους. Παρακαλώ λοιπόν αυτοί που ασχολούνται με το θέμα της Ουκρανίας ε, να καταλάβουν τη σημασία της χώρας και να ετοιμάσουν ένα δημοσιονομικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της υποδομής στα σύνορα μεταξύ Ουγγαρίας ε, και Ουκρανίας για τη διευκόλυνση της ε, εισόδου των Ουκρανών αυτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης και σε σχέση με την μεταναστευτική κρίση και τα τρομοκρατικά πλήγματα. Πρέπει να δούμε την ε, λήψη μέτρων για την ε, διασφάλιση της ε, ασφάλειας της ποιότητας. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από δύο χρόνια εξουσίας, ανάληψης εξουσίας δεν έχει καταλήξει στις ε, πιο σωστές πολιτικές. Πώς θα βελτιωθεί η εμπιστοσύνη, το κλίμα εμπιστοσύνη των πολιτών σε σχέση με την Ευρώπη λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα και καμιά θετική αλλαγή στη ζωή των πολιτικών και πρέπει εδώ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ληφθούν υπόψη οι ρήτρε ε, της συνθήκες για την ασφάλεια και την ε, ποιότητα ζωής ε, των πολιτών. Δεν μπορούμε να υπαρκεστούμε με τίποτα άλλο. Οι πολίτες απαιτούν μια αλλαγή και στην επικοινωνία. Ευχαριστώ. <laughs> Πηγαίνετε πάρα πολύ γρήγορα και δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Ο κύριο Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την απόφαση που ελήφθη για το Brexit. Ακούγοντας κάποιους από τους συναδέλφους εδώ, νιώθουν ότι το ίδιο που συνέβη πριν από 25 χρόνια. Πριν από την διάλυση της Ιουκοσλαβίας θα μπορούσε το Brexit να είναι ένας πρόλογος στην διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να συμβεί εγώ προσωπικά βέβαια. Θα ήθελα να μιλήσουμε για καλύτερους δεσμούς ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να είναι πιο ρόδινο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως δυστυχώς να αλλάξει η πολιτική μας, γιατί αν συνεχίσουμε θα διαλυθούμε. Benito ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στο, στο Καλέ είναι πραγματικά επέσχυντη. Έξι μήνες μετά τις τελευταίες ε, εξώσεις ο πληθυσμό αυξήθηκε πάνω από 3.000 ενώ η έκταση μειώθηκε σημαντικά επιδεινώνοντας τις, ε, την κατάσταση. Δίπλα στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει Α, ένα τείχος ε, προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ. Το, η εικόνα της Ευρώπης ε, Φρούει, Από τη μια μεριά η αθλειότητα των προσφύγων που προσπαθούν να φύγουν από τον πόλεμο και από την άλλη η βίαιη απάντηση των δυνάμεων της ασφάλειας. Όλα αυτά για να δημιουργηθεί μια εικόνα δυναμίας διαχείρισης τελείως ψευδής. Η εντύπωση αυτή της εισβολής που αρέσει τόσο στην δεξιά είτε ακραία είτε λαϊκιστική. Θα πρέπει να υποδεχθούμε τους ανθρώπους με δικαιώματα όταν το χρειάζονται. Αυτό ε, ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αλλάξει. Θα έχουμε χιλιάδες ε, πρόσφυγες. Ο κύριος Καμπράς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χτες, 11 Σεπτεμβρίου του 2016, ένα εκατομμύριο άτομα σχεδόν βγήκαν στους δρόμους της Καταλωνίας για να γιορτάσουν την εθνική τους γιορτή, ζητώντας την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Αυτό έγινε χθες. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά δεν υπήρξε στην Ευρώπη τόσο μεγάλη κραυγή όπως αυτή που ακούγεται στη χώρα μου. Ωστόσο η Ισπανική κυβέρνηση αντίθετα από οποιαδήποτε δημοκρατική λογική αρνείται να κάνει να διεξάγει ένα δημον ψηφίσμα όπως έγινε στην Σκοτία, ούτως ώστε όλος ο κόσμος να γνωρίζει αν η βούληση ανεξαρτησίας είναι πλειοψηφική ή όχι στην Καταλωνία. Σήμερα θέλω να καταγγείλω εκ νέου στο Κοινοβούλιο την αντιδημοκρατική άρνηση των Ισπανικών αρχών. Σε μία δημοκρατία δεν χρησιμοποιείται ο νόμος για να φημώσουμε την ελευθερία. Σε μια δημοκρατία ο νόμος είναι η βούληση του λαού. Στην Ισπανία αυτό ξεχάστηκε. Στην Καταλωνία το θυμόμαστε και το απαιτούμε. Ευχαριστώ. Κυρία Μάλιστα κυρία Πρόεδρε. Κανείς δεν έμαθε από τόσα συνέβησαν η γερμανική κυβέρνηση και η Γαλλία καταλήγουν στην εξαιρετική ιδέα λέει να δημιουργηθούν στρατεύματα ευρωπαϊκά με κονδύλια ευρωπαϊκά δηλαδή με τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και για τα ελάχιστα έσοδα θα διατεθούν χρήματα για αυτούς τους σκοπούς δηλαδή και δεν φτάνει το ότι ζητείτε να έχουν πόρους τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισφορές ε, και τέλει, αλλά το να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει σε αυτό τον τομέα. Κυρίες και κύριοι, οι Βρετανοί ούτε με το ένα πόδι δεν βρίσκονται εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και υπάρχουν σκέψεις ε, να υλοποιηθούν τέτοια μέτρα φαίνεται ότι δεν έχουν μάθει κάποιοι και ούτε θέλουν να μάθουν και να συναγάγουν τα σωστά συμπεράσματα. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα οι πολίτες μας και τα δημοψηφίσματα θα το καταδείξουν αυτό. Ο κύριος Πολτσακ. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο αφορά την ολοφορία έκφρασης ή τις προσωπικές ελευθερίες στη Γαλλία. Να αναφερθώ στα Μπουρκίνη δεν ομιλώ σαν ένας βουλευτής, αλλά σαν ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος θέλει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά δεν θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον είναι καθαρά εσωτερικά θέματα. Εμείς θα πρέπει να ασχοληθούμε μετά τα της και τίποτα περισσότερο. Δεν πρέπει να είμαστε κατά της αρχής της επικουρικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τη βούληση των λαών και των κυβερνήσεων. Θα πρέπει να υποστηρίζει τους πολίτες σε σχέση με αυτά τα οποία επιθυμούν. για δεκαετίες, λέει η κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ, δίνει εκατομμύρια στην βόρειο-ανατολική Ευρώπη, την περιοχή από όπου εκλέγομαι. Τα τελευταία χρόνια περιμένουμε ε, σχεδόν μισό δις ε, στην σύνολη περιοχή, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας, προωθώντας την καινοτομία και την αριστεία. Μετά το Brexit, δυστυχώς μία από τις πιο φτωχές περιοχές της ε, Ένωσης θα γίνει ακόμα πιο φτωχή. Μα έλεγαν αυτοί που ήταν υπέρ της αναχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας ότι το Brexit θα μας ωφελούσε οικονομικά. Αλλά δυστυχώς ε, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι πραγματικότητα. Ζητώ από τη Βρετανική κυβέρνηση έτσι ώστε όλα τα χρήματα που έχουν ε, γίνει αντικείμενο υπόσχεσης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν στην περιοχή μου. E η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η κυρία Χάρκιν, θεωρεί ότι πρέπει να περιμένει η Ιρλανδία να εισπράξει απλά 13 δις, να τα ξοδέψει σε νοσοκομεία, σε σχολεία. Ωστόσο σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ετοιμάζονται να φάνε το κομματάκι από την πίτα. Αυτό που θα μείνει στην Ιρλανδία είναι πολύ λίγα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί η Βρυξέλλε, να χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για να κορυδεύουν τους Ιρλανδούς. Δεν τα κέρδισαν αυτά οι Ιρλανδοί. Η ίδια επιτροπή ωστόσο είναι αυτή που είναι μέλος της Τρόικας που μας υποχρέωσε να καλύψουμε 60% περίπου του κόστους της ε, κρίσεως και να πληρώσουμε κάποιους ε, ιδιοκτήτες, κάποιους μετόχους τραπεζών. Η ΤΡΑ, η Επιτροπή είναι αυτή που υποσχέθηκε 350 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα ε, εάν δεν, ε, δεν ψηφίσουν να φύγουν. Αυτό είναι πραγματικά παράδεκτο από πλευρά τη επιτροπή. Μα, ο κύριο Κάρθη. Πρόεδρε, η απάντηση της τότε κυβέρνησης του Φίνεφόλ στην τραπεζική κρίση και σε πυλώνες όπως την, ε, το βάρος του ιδιωτικού χρέους της οικογένεια και η επιβολή της σκληρής λιπτότητας ήταν ε, ε, μία από τις ε, πλευρές της κρίσης. Η άλλη ήταν η δημιουργία του ΝΑΜΑ, του National Asset Management Agency. είναι σαφές το ότι η πώληση του ΝΑΜΑ το 2014 στην Βόρεια Ιρλανδία έγινε μετά από διαφθορά πουλήθηκαν σε ταμεία όρνεα σε πολύ χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Όλες οι πωλήσει, ε, όλες οι συναλλαγές του ΝΑΜΑ πρέπει να ανασταλούν αμέσω. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση της Λαδία δεν μπορεί να καλέσει, δεν μπορεί να αγνοήσει την ανάγκη να υπάρξει μια εξεταστική επιτροπή για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμα. Η έρευνα πρέπει να καλύψει πώς δημιουργήθηκε αυτή η απάτη. Ευχαριστώ. Κύριος Πάβελ. Υπάρχουν πολλές απειλές για τους λαούς της Ευρώπης, οι κλιματολογικές αλλαγές. Being Υπάρχουν τα προβλήματα βέβαια με διάφορα παράσιτα στην φυτική παραγωγή. Ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν στο νότο της ε, Ιταλίας είναι ένα ζωήφιο, μια άκαρηση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό θα πρέπει ε, να απαγορευτεί η εξαγωγή τέτοιων προϊόντων γιατί αλλιώς φοβάμαι ότι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα στην ε, ε, παραγωγή μελιού σε όλες τις περιοχές της υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις ψηφοφορίες ψηφοφορίες ή για τις εκλογές καλύτερα σε σχέση με την ανάδειξη του Κοινοβουλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, ε, όχι μόνο θα διεξαχθούν στην επικράτεια της Ρωσίας αυτές οι εκλογές αλλά και στην ίδια την Κρυμαία που προσαρτήθηκε από την Ρωσία. Το Κρεμλίνο θέλει να νομιμοποιήσει λοιπόν αυτές τις εκλογές στην Κρυμαία επικαλούμενο το δημοψήφισμα του Μαρτίου 2014. Όμως όλα αυτά αντιβαίνουν την απόφαση 68-62 ε, των Ηνωμένων Εθνών και η Κρυμαία αποτελεί από, ε, άρρηκτα τμήμα της ε, Ουκρανίας. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης από πλευράς της Ρωσίας και παραβίασης ε, και καταπάτησης του διεθνούς δικαίου από την Ρωσία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τανασέσκου. Ευχαριστώ Συνάδελφοι, η, η ολοκλήρωση της ε, ε, η αύξηση των εισόδων δημιουργεί σοβαρές ε, ανησυχίες στους εταίρους εκτός Ένωσης, ιδίως στους εταίρους μας μετά την, έξοδο, μετά την πιθανότητα έκδοση της Βρετανίας στην Ιαπωνία υπάρχει μια επιφυλακτικότητα για τις επενδύσεις ε, της Ιαπωνίας στη Βρετανία. Αυτό έχει επιπτώσει στο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Φαρμάκων που βρίσκεται εκεί. Ίσως θα ήταν λοιπόν να ξανασκεφτούμε τον ενδεχόμενο να αλλάξουμε την έδρα της Υπηρεσίας Φαρμάκων. Ε, είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να πάρουμε μια σχετική απόφαση, γιατί αν η Μεγάλη Βρετανία δεν παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί μια υπηρεσία της Ένωσης να βρίσκεται εκεί. Η Ρουμανία έχει μια μεγάλη παράδοση, έχει σαφή ιστορικό, σαφές ιστορικό μελετών στον τομέα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να δείξει μεταξύ άλλων ότι θέλει να δουλέψει υπό μια αλληλέγγυη Ευρώπη στην οποία όλα τα κράτη-μέλη έχουν ισότιμο ρόλο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι εγώ, λέει εγώ είμαι. Ποια είναι αυτή. Η κυρία Άντερσον, η επιβρετανική κυβέρνηση, προσπαθεί να μας κρατήσει στο σκοτάδι και τις προθέσεις που έχει ως προς το μέλλον, δημιουργώντας ε, αβεβαιότητα για το τι σημαίνει το Brexit για τους λαούς της Σκοτίας, ε, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Ουαλίας. Ο κόσμος δεν ξέρει και αυτό ε, πλήττει και τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινότητες. Η Βρετανική, κυβέρνηση, η Βρετανική κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει τρόπους με τους οποίους η δημοκρατική βούληση του Βορρά θα της Βόρειας Ιρλανδίας θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Το 56% ψήφισαν υπέρ του Remain υπάρχουν μια σειρά ανθρώπων ε, που, που ζητούν κάτι τέτοιο και που σαφώς τονίζουν ότι το remain σημαίνει remain. Εκατοντάδες χιλιάδες Βορειοϊρλανδών έχουν Ιρλανδικά διαβατήρια που σημαίνει ότι είναι πολίτες της Ένωσης. Για το λόγο αυτό το remain που ψηφίσαμε πρέπει να είναι πραγματικό remain. Ο κύριος Τσάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια οντότητα για την οποία διεξήχθη μια συζήτηση για τις ε, μειονότητες όπου ο κύριος Τίμερμανς είπε θα εκπονηθεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση και την επίλυση των προβλημάτων. Αξιολόγησε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα αυτό το πρόγραμμα, όπως και η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πέρυσι, αυτό το πρόγραμμα παίρνει ένα εκατομμύριο ευρώ. Αποκαλείται Ευρώπη Ενωμένη στην Πολυμορφία και σε σχέση με τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο θα υπάρχουν λέει οι αυτές οι δράσεις μέχρι σήμερα δεν έγινε όμως τίποτα είναι απαράδεκτο αυτό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να το τονίσω και πάλι αν από τον Οκτώβριο δεν, έχει, δεν γίνει κάτι θα απευθυνθώ στα μέσα ενημέρωσης Νεγκρέσκου παρακαλώ στο σήμερα πάμε όλα παιδιά επιστρέφουν στα σχολεία τους και διαρωτώμεθα η εκπαίδευση θα παρέχει ένα καλύτερο πλαίσιο για το μέλλον των παιδιών. Θεωρείται δαπάνη η εκπαίδευση, όμως είναι επένδυση στο μέλλον και στη ζωή των παιδιών. Αυτή η προσέγγιση κάνει τους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα στους αριθμούς και στα λογιστικά και όχι στη ζωή των παιδιών και παγιδεύονται στα γραφειοκρατικά ζητήματα και δεν επικεντρώνονται στην ουσία. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά πρότεινε μέτρα προσπαθώντας να πείσουν τους νομοθέτες ότι θα πρέπει να αναλυθεί συνεκτική δράση για την υποστήριξη αυτών των μέτρων. Ως νέος Ευρωβουλευτής πρέπει να πω ότι σήμερα οι Ρουμάνοι ναι, νέοι, στη Ρουμανία επιθυμούν πραγματικά να είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ντέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε στόχος των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων είναι να ενταχθούν στην, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επί πολλά χρόνια αυτό ε, δεν λύθη υπόψη. Χαίρομαι για το ότι βλέπω ότι το ΕΛΚ εργάζεται ενεργά προς όφελος αυτών των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Οι χριστιανικές και δημοκρατικές αξίες έχουν τεράστια αξία και σε σχέση με την, ε, τις εκλογές και στην ε, ε, Κροατία και στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν και στη Μακεδονία και στην Βοσνία Ζεγοβίνη λέει ο μιλητής ιδιαίτερα για τη Βοσνία Ζεγοβίνη που θέλει να γίνει ένα συνδεδεμένο συνδεδεμένος εταίρος, συνδεδεμένο κράτος μέλος Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτές τις φιλοδοξίες που θα συνεισφέρουν στο να σταθεροποιηθεί η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαΐτοβα κλείνει. Συνάδελφοι, θέλω να μιλήσω για να τονίσω την, ε, τις εντάσεις που αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία. Ήμουν μέλος του ΕΜΠΛ και είχα υποτίθεται πήγαινα την άλλη εβδομάδα σε μια αποστολή στην Τουρκία η οποία ακυρώθηκε λόγω της τρέχουσας ε, κατάστασης ε, όπου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, δεν είναι βέβαια η ασφάλειά μας και δεν θα μπορέσουμε να επισκεφθούμε μια σειρά θεσμικών οργάνων. Αυτό με ανησυχεί. Η Τουρκία απαιτεί απελευθέρωση των θεωρήσεων. Εγώ ωστόσο ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση στη χώρα και θα ήθελα να γίνεται σεβαστή συμφωνία Ένωσης Τουρκίας και από πλευράς Τουρκίας. Ωστόσο, εάν ε, η, μετα... η μετακίνηση στην Τουρκία, ωστόσο, δημιουργεί αβεβαιότητες γιατί ε, δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο στις 9. Υπάρχει ημερήσια διάταξη στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Διακόπτη συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.